Καλημέρα σας. Ξεπεράσαμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας, η οποία είναι και διάσκεψη ουσιαστικά. Έχουμε προσκαλέσει επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, από πανεπιστήμια και από άλλα ερευνητικά κέντρα. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θα ακούσουμε λοιπόν σήμερα και να ξεκινήσουμε. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να εγκρίνουμε την ημερήσια καταξία όσο έχει. Έχουμε τη σε 20 γλώσσες εκτός από τσεχικά, σλοβακικά, και γαλλικά. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και ας κοιτάξουμε τώρα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Της 7ης Ιανουαρίου συγκεκριμένα. Και της 11 η Ιανουαρίου. Και τα πρακτικά του Ιουνίου δεν είχαμε ε, εγκρίνει. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούνται εγκεκριμένα λοιπόν τα πρακτικά. Τώρα, κάποια στοιχεία για το περιεχόμενο. Για το βασικό σημείο της συνεδρίασής μας. Θα ακούσουμε μια ανάλυση για την γεωργική πολιτική παγκοσμίω, μαθήματα για την περιοδική κοινή γεωργική πολιτική Θα ακούσουμε την Σιμών Στερλή και τον Ραέλ Γιόμινελ. Εμπειρογνώμονες τους οποίους γνωρίζουμε καλά. Και οι συντονιστές αποφάσισαν στην προηγούμενη συνεδρίασή τους να δοθεί εντολή για την διεξαγωγή της ε, μελέτης αυτής στις 22 Νοεμβρίου 2017, γιατί θέλουμε να έχουμε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τους ε, εμπορικού μας εταίρους στην Ιαπωνία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το καθεξής, για να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε την όλη πολιτική. Το θεματικό τμήμα βοήθησε επίση με τη σειρά του και σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις ε, πτυχές ε, των οριζοντίων σχεδίων, ε, των στρατηγικών σχεδίων μάλλον, τη οριζόντια, του οριζόντιου κανονισμού για την κοινή οργάνωση τη αγορά. Όπω γνωρίζετε, εργαζόμαστε επί των τριών αυτών νομικών εγγράφων και Ελπίζουμε να μην έχουμε καθυστερήσει ήδη σε ό,τι αφορά τη μελέτη αυτή. Σε κάθε περίπτωση θα μας βοηθήσει η μελέτη αυτή, η έρευνα αυτή, να κατανοήσουμε σε βάθος την κοινή γεωργική πολιτική για να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε και μακροπρόθεσμα την γεωργική πολιτική. Με την υποστήριξη και τρίτων χωρών. Να ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση. Χαιρόμαστε λοιπόν που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Έχουμε προγραμματίσει και λίγο χρόνο για την παρουσίασή σας. Και φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετό χρόνο ομιλία. Νομίζω ότι 15 λεπτά είναι ρεαλιστικό διάστημα. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την συνεδρία. Χαίρομαστε ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε αυτή την συγκεκριμένη μελέτη. Είμαι από το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης και έρευνα, αλλά συνεργαστήκαμε στενά με μια ομάδα από ένα ερευνητικό κέντρο και πανεπιστήμιο ε, όπου συνεργαστήκαμε με τον Ρόελ και δεν ήμασταν οι μόνοι, ήταν και άλλοι δύο που συνεργάστηκαν στενά, Χόλγα Πάπστα και Χουπ Σίλβης. Σε πέντε χώρες έχουμε εστιάσει όπως θα δείτε. Συνεργαστήκαμε στενά με ειδικού, ε, Τζεφ Κόνορ από την Αυστραλία, David Freshwater από τη ΣΥΠΑ, Μίκη Τάρο Σομπαγιάση και Γιούκη Οκονοσίτα από την ε, Ιαπωνία και, και Σφανκότερα από τον Καναδά. And we had Alexander Και Αλεξάνδερ Τσόν από την Ελβετία. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν Αυτό που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τώρα, είναι συντομία καταρχάς η προσέγγιση για τη μελέτη αυτή που ακολουθήσαμε, ποιος ήταν ο στόχος και εν συνεχεία θα δούμε πώς εξελίσσεται γενικά η γεωργική πολιτική, ποιες ήταν οι βασικές τάσεις, ε, καινοτομίε ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα παρουσιάσουμε έπειτα τις ε, μελέτες χωρών με μια σύντομη παρουσίαση για την κάθε χώρα. Επίσης θα σας παρουσιάσουμε μόνο λίγα μέσα, μόνο λίγα εργαλεία, γιατί δεν ε, νομίζω έχουμε χρόνο να ψέλθουμε σε λεπτομέρειες για όλα αυτά. Θα σας πούμε τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και βεβαίως θα κάνουμε προτάσεις πολιτικής και συστάσεις. Ο στόχος της μελέτης ήταν να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής από τη συγκριτική ανάλυση των γεωργικών πολιτικών άλλων χωρών. να βοηθήσουμε και για τη χάραξη πολιτικής μέσω της ε, συλλογής γνώσεων και για να βελτιωθεί και η κοινή πολιτική όχι μόνο άμεσα αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα. Ο στόχος μας δεν ήταν μόνο να μελετήσουμε τα διάφορα εργαλεία αλλά και σε επίπεδο υποστήριξης ε, που παρέχεται να δούμε τι γίνεται. Στη μελέτη λοιπόν εξετάσαμε τις παγκόσμιες τάσεις σε επίπεδο στατιστικών δικτών του ΟΣΑ, τις τάσεις και τις πρόσφατες αλλαγές, νέες καινοτομίες και στη βιβλιογραφία και διανοήσαμε πέντε αναλυτικές μελέτες χωρών, τις οποίες επιλέξαμε Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Ελβετία, ΗΠΑ είναι πέντε χώρες τις οποίες επιλέξαμε διότι είναι παγκόσμια ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ένα διαφορετικό επίπεδο υποστήριξη. Άλλες χώρες υψηλότατο επίπεδο στήριξη στη γεωργία και άλλες χώρες με πολύ χαμηλό. Επίσης, ε, είδαμε ενδιαφέροντα προγράμματα στήριξης, ε, μελετήσαμε τις ομοιότητες ε, ε, των πολιτικών των χωρών αυτών με την κύλη πολιτική. Σε άλλες χώρες υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες, σε άλλες καθόλου. Και είδαμε τα θέματα της ασφάλειας τροφίμων. Μιλήσαμε δηλαδή για χώρες ε, που εισάγουν βασικά γεωργικά προϊόντα. Δέκα κράτη-μέλη επίσης μας έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές για τη γεωρική πολιτική. You want to continue? So the, the, the first uh, topic is Το πρώτο λοιπόν θέμα είναι η ε, εξέλιξη της ε, γεωργικής πολιτικής και αν δείτε τη μελέτη, βλέπετε ότι υπάρχει μία σύνθεση ζητημάτων, αλλά αν δούμε τους στόχους υπάρχουν ομοιότητες. Είδαμε όλες τις ε, χώρες, κατά πόσο υπάρχει περιορισμός των πόρων και βλέπετε και περιβαλλοντικές ανησυχίες, ιδιαίτερα τις κλιματικές αλλαγές και φυσικά και τη μελλοντική ζήτηση σε τρόφιμα, όπου θα πρέπει να προτρέξουμε. Γι' αυτό θέλουμε να προωθήσουμε την οικονομική βιωσιμότητα καθώς και την αποδοτική χρήση των πόρων. Αν δούμε τις δύο τελευταίες δεκαετίες, και αν δείτε την στήριξη αυτών των χωρών, βλέπετε τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ως προς το συνολικό επίπεδο υποστήριξης. Αλλά η σύσταση, η σύνθεση της υποστήριξης έχει αλλάξει. Αν δείτε τις αναδυόμενες οικονομίες, δηλαδή αν δούμε την Κίνα Πρωταρχικά βλέπετε ότι υπάρχει υποστήριξη, η υποστήριξη των τιμών αγοράς από τον ΩΣΑ. Και είναι το ίδιο με αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν, δηλαδή στήριξη τιμών ε, που οδηγεί σε στρέβλωση δηλαδή οδηγεί σε στρέβλωση τιμών αγοράς και δίνει λανθασμένα μηνύματα. Στις χώρες του Όσα, βλέπετε ότι υπάρχει μία αλλαγή. Δηλαδή μειώνεται η υποστήριξη, η στήριξη αυτή στις τιμές αγοράς και βλέπετε ότι από το 2000 και μετά υπάρχουν καθαρά περιβαλλοντικά μελήματα και περισσότερα μέσα και καταβολές για περιβαλλοντικούς σκοπούς για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους και μετά το 2010 σε μερικές χώρες και νωρίτερα υπάρχει και η διαχείριση κινδύνων που κατέχει υψηλότερη θέση. Αυτό αφορά και τις χώρες του όσα έχουμε άμεσες καταβολές, λιγότερη υποστήριξη τιμών αγοράς και βεβαίως ε, πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων. Και αν δείτε την συνολική υποστήριξη, το 70% φτάνει στους παραγωγούς, στην υποστήριξη παραγωγών. Και αν θέλετε να δείτε πώς έχει σε σχέση με την ε, συνολική αξία παραγωγής φτάνει στο 18%. Δηλαδή μείωση κατά 40% σε σχέση με την αρχή της περίοδου. Έχουμε λοιπόν μία μείωση και παράλληλα αυξάνεται και η γεωργική παραγωγή. Αν και η στήριξη λοιπόν είναι σταθερή, η παραγωγή έχει ε, αυξηθεί. Άρα ε, ο δείκτης αναμονάδα είναι πιο χαμηλός. Και αν δείτε τις αγορατικές υπηρεσίες, μιλάμε για ένα 80% του συνολικού εισοδήματος, το οποίο δεν είναι, δεν είναι κάτι το ουσιαστικό δείτε τις γενικές υπηρεσίες τον ε, τομέα της τεχνογνωσίας ή καινοτομίας και διάδοση της γνώσης στους ε, αγορότες, βλέπετε αυτό ανέρχεται στο 20% του ε, τιμολογίου, θα μπορούσαμε να πούμε, υποστήριξης. Εάν το συνδέσετε με επιχειρήσεις εκτός γεωργίας, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις ε, που να δίνει το 20% στην έρευνα και την ανάπτυξη, να αποδίδει δηλαδή τόσο υψηλό ποσοστό. Εδώ βλέπετε την εξέλιξη στήριξης αναχώρα ως ποσοστή αναλογία του ΑΕΠ. Και βλέπετε ότι το 1% του ΑΕΠ καταβάλλεται στις, ε, στη γεωργική στήριξη. Στην Αυστραλία πολύ χαμηλός ο δείκτης, ο Καναδάς είναι πιο ψηλά, η Ελβετία έχει τον υψηλότερο δείκτη. Βλέπετε δύο δείκτες για την αρχή 95-97 ενώ ο μπλε δείκτης αφορά τα πρόσφατα χρόνια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία ουσιαστική μείωση ως ποσοστία αναλογία επί του ΑΕΠ, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη του, στο γεωργικό τομέα. Ας ε, στρέψουμε την προσοχή μας στις χώρες. Η Αυστραλία έχει την χαμηλότερη υποστήριξη, όπως και η Νέα Ζηλανδία. Και χορηγούνται, ε, μάλλον χρηματοδοτούνται οι έρευνες σε σχέση με την ξηρασία, ας πούμε, στην Αυστραλία. Στον Καναδά, Ένα στόχος είναι η προστασία της γεωργίας από την γενικότερη φύση που περιβάλλει τη χώρα, αλλά το κόστος θα πρέπει να είναι χαμηλότερο και γι' αυτό ο Καναδάς ελέγχει την παραγωγή με, την, με σχέδια διαχείρισης και αυτό αφορά τα γαλακτοκομικά, τα πουλερικά, ενώ οι καταναλωτές καταβάλουν υψηλότερο τίμημα υποστηρίζοντας τους αγρότες. Στον Καναδά προσδίδουν μεγάλη σημασία και στη διαχείριση κινδύνου για να βοηθήσουν τους αγρότες σε αυτό το τομέα. Στην Ιαπωνία υπάρχει θέμα ε, αυτοδυναμίας, αυτοδυναμίας ιδιαίτερα στον τομέα του ρυζιού έτσι ώστε να υπάρχει αυτάρκεια και να υποστηριχθούν οι αγρότες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι η γεωργική εκμετάλλευση είναι πολύ μικρή, 1,5 εκτάριο όσον αφορά τους οριζόνες. Και υπάρχει και το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού, γιατί ο μέσος αγρότης είναι 70 χρονών. Και Άρα διαφέρει ε, από το μέσο όρο. Στην, ε, στην Ελβετία, συγγνώμη, high level of price In that sense are a Στην κατάσταση, η κατάσταση είναι παρόμοια με την Ιαπωνία. Και εδώ ε, έχετε ένα αναπτυγμένο σύστημα άμεσων πληρωμών, όπως ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. για την υποστήριξη της γεωργίας σε μειονεκτούσες περιοχές και την παροχή αγαθών προς την, τις κοινότητες αυτές. Γι' αυτό υπάρχουν και οι άμεσες πληρωμές, η άμεση στήριξη στις ΕΠΑ. Βλέπετε ότι υπάρχει επιδότηση της γεωργίας υψηλή επιδότηση σε αντίθεση με την Ελβετία που έχουν και κυκλικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν είναι χαμηλές οι τιμές, οι γεωρικές τιμές, τότε η υποστήριξη είναι υψηλή. Υπάρχει δηλαδή στοχοθέτηση με βάση τις συνθήκες της αγοράς. Τώρα να κοιτάξουμε λοιπόν σε πιο πολλές λεπτομέρειες σε τις ε, συγκεκριμένες υποθέσεις και περιπτώσεις. Καταρχά, τι έκαναν οι εμπειρογνώμονε αναχώρα. Ζητήσαμε να μα δώσουν μία επισκόπηση των στόχων ε, αναχώρα και να δούμε τι πρόσφατε ε, τάσει πέρα από τι οικονομικέ τάσει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ανάπτυξη των εργαλείων. Ζητήσαμε λοιπόν να μας δώσουν ένα μακρύ κατάλογο εργαλείων για στόχους ε, παρόμοιους με αυτούς που έχουμε στην ΚΑΠ σήμερα. Λάβαμε λοιπόν 75 μέσα, μέτρα που σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με τους στόχους της ΚΑΠ και ζητήσαμε να κοιτάξουμε βασικά εργαλεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα φάση στην ΚΑΠ και εργαλεία τα οποία διαφέρουν, διαφέρουν σημαντικά από αυτά που εφαρμόζουμε σήμερα στην ΚΑΠ. Και άρα καταρτήσαμε μια λίστα, ένα κατάλογο 75 εργαλείων, εκ των οποίων διαλέξαμε 70 για ανάλυση σε βάθος. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν ένα πίνακα για τον αντίκτυπο των ε, μέτρων αυτών, ένα πλαίσιο για να υπάρχει συγκρισιμότητα και προσμέτρηση του αντικτύπου των μέτρων και να μας βοηθήσει γενικά στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τι εξετάσαμε, λοιπόν. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Εργαλεία για το περιβάλλον, για το κλίμα. Αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο όγκο των πληροφοριών στην μελέτη, αλλά και μέτρα ανάπτυξης ε, της υπέτρου. Δεν είδαμε πολλά που να είναι ενδιαφέροντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέτρα για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και μέσα για καινοτομία. Αλλά αυτά τα μέσα είχαν άλλον έναν βασικό στόχο και στοιχεία, αν θέλετε, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καινοτομία και στην γνώση. Αυτά ουσιαστικά είναι πιο ενσωματωμένα σε, από άλλους ε, τομείς. Είχαμε και μέτρα marketing και μέτρα για τις εγγύησεις. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησαμε για την εκτίμηση, την αξιολόγηση των μέτρων είναι κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αξιολόγηση. Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνοχή, για παράδειγμα, προσθέσαμε και κάποια κριτήρια τα οποία θεωρούσαμε ότι ήταν ενδιαφέροντα ή σημαντικά σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη συμβατότητα, το πόσο εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο σε μια ευρωπαϊκή επιχειρήση, σε ένα ευρωπαϊκό αγρόκτημα και πώς μπορεί ένα τέτοιο μέτρο να συμβάλλει και σε άλλους στόχους ΚΑΠ, πέρα από αυτούς που περιγράφαμε. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να κοιτάξουμε και τα 17 αυτά εργαλεία, τα οποία προφανώς ε, περιλαμβάνονται στην έκθεση για την ε, μελέτη και την έρευνα. Θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα για την ε, προβλητική ανάπτυξη, για την διαχείριση κινδύνου και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ένα από τον κάθε τομέα. Καταρχάς λοιπόν ο στόχος της ε, μείωσης της επίπτωσης ε, στο κλίμα. Εδώ βλέπετε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. για τη μείωση εκπομπών άνθρακα. Αυτό δεν είναι τμήμα της ε, γεωργικής πολιτικής, είναι μάλλον τμήμα της πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος, για το περιβάλλον. και ουσιαστικά χρησιμοποιείται στην Αυστραλία για την ε, επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον. Και το εργαλείο, το μέσο αυτό χρησιμοποιείται μέσω αντίστροφου πληστηριασμού. Άρα, οι αγρότες εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για το μέτρο αυτό, βάζουν μια τιμή, ορίζουν μια τιμή και ουσιαστικά το καλύτερο, η καλύτερη απόδοση τα χρήματα αυτά τελικά είναι αυτή που χρηματοδοτείται. Τα τελευταία χρόνια περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν με τον τρόπο αυτό και τα πιο πολλά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν είχαν να κάνουν με την, τον καθαρισμό περιοχών, την αφαίρεση επίσης ε, ζώων από κάποιες περιοχές. Ε, ο αντίκτυπος τώρα. Η αποτελεσματικότητα και η αποφατικότητα είναι μάλλον μέτρια, διαπιστώσαμε, αλλά σε επίπεδο αγροκτήματος είναι συμβατό το μέτρο αυτό. Είναι ένα εύκολο μέτρο να εφαρμοστεί δηλαδή σε επίπεδο αγροκτήματος. Και επίσης πολύ συμβατό με άλλους στόχους που χρηματοδοτούνται. Το δεύτερο το εργαλείο που κοιτάξαμε και το οποίο θέλουμε να σας παρουσιάσουμε με μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρεια, είναι ένα μέτρο που αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Εδώ πρέπει να σα πω ότι εξετάσαμε διάφορα τέτοια μέτρα για τη διαχείριση κινδύνου. Μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε σε δύο κατηγορίε. Καταρχά ε, περιορισμό κινδύνου και το άλλο είναι η μεταφορά κινδύνου. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την πρώτη κατηγορία ε, περιορισμό του κινδύνου για να περιορίσουμε κάποιου απλού κινδύνου ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διακύμανση τιμών. Πρόκειται για χαμηλού κόστου μέτρο. Εξετάσαμε το πρόγραμμα Angrill Invest του Καναδά. Ο στόχο είναι να σταθεροποιηθούν τα εισοδήματα των γεωργών. Πρόκειται για ένα σύστημα αμα, λογαριασμού ταμιευτηρίου, το οποίο το διαχειρίζονται οι συμμετέχουσες τράπεζες τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στους λογαριασμούς αυτούς, τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο ποσοστό. είναι συμβατό με τη διαχείριση τέτοιων κινδύνων. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του ως μέτρο. Αλλά είναι ουσιαστικά μόνο εν μέρη συμβατό με τους άλλους στόχους της ΚΑΠ. Το τρίτο μέτρο το οποίο εξετάζουμε είναι ένα μέτρο που υπάρχει στην κατηγορία για την ανάπτυξη της υπέτρου. Όπως σας είπα, δεν ήταν πολλά τα καινοτομικά εργαλεία τα οποία να διαφέρουν από τα μέτρα ανάπτυξη της υπέτρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί ουσιαστικά η πολιτική για την ανάπτυξη τη υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει μια ευρία γκάμα μέτρων που δεν χρησιμοποιούνται πουθενά άλλου στον κόσμο. Είδαμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο εφαρμογής για τέτοια μέτρα. Ένα παράδειγμα λοιπόν που κοιτάξαμε Στην Ιαπωνία έχουμε την πληρωμή πολυλειτουργικότητας. Ο στόχος λοιπόν του μέτρου αυτού είναι να διατηρηθεί ή να ανοικοδομηθεί η υποδομή στην Ήπετρο. Δρόμοι, άρδρευση και η διαμόρφωση του τοπίου της Ήπετρου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα οι πόροι αυτοί καταβάλλονται σε οργανώσεις, ενώσεις για όχι σε άτομα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτό όντως προωθεί και την κοινωνική συμπερίληψη και δίνει μια σύνδεση μεταξύ της ε, γεωργικής κοινότητας και της μη γεωργικής κοινότητας στην Ήπεθρο. Επίσης, ε, προωθεί και άλλους στόχους της κάπο όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση υδάτων. Αλλά, φυσικά, ο απότερος στόχος του μέτρου αυτού δεν εντάσσεται ουσιαστικά στο πλαίσιο της ΚΑΠ, γιατί είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα το οποίο προωθεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεγάλης έκτασης. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι πολύ μικρή κλίμακα στην Ιαπωνία, άρα υπάρχει αυτή η τάση να υποστηρίζονται μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Η αποτελεσματικότητα τώρα του μέτρου αυτού. Θεωρήσαμε ότι είναι μάλλον περιορισμένη. Γιατί ουσιαστικά χρηματοδοτεί την συντήρηση. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να γίνεται. Τα έξοδα ουσιαστικά για την καλλιέργεια τα αναλαμβάνει ο Γιώργος. αλλά η συμβατότητα είναι υψηλή και η συνοχή είναι υψηλή και μόνο και μόνο ο τρόπος εφαρμογής αποτελεί ένα ενδιαφέρον μέτρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω λοιπόν το λόγο τώρα πάλι στον συνάδελφο για να συνοψίσει τι συστάσει μας. Ωραία. Να συνοψίσουμε λοιπόν τις συστάσεις μας. Πρώτη παρατήρηση. Αν γίνει σύγκριση Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλε χώρε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε προχωρημένη θέση στη γεωργική πολιτική με ένα συνολικό ε, στόχο ε, πολιτικών και έχει και στη διάθεσή της μέσα, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να διδαχθεί πράγματα από τις άλλες χώρες. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων, έχουμε την εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνων φυσικά στην κοινή γεωργική πότη και όπως είπε η Σιμών, με δύο τρόπους μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Να τον συγκρατήσει σε επίπεδο αγροκτήματος ή να τον μεταφέρει σε τρίτο μέρος, σε κάποιον τρίτο. Αυτό το οποίο θεωρήσαμε ενδιαφέρον από το καναδικό και το αυστραλιανό παράδειγμα κυρίως, είναι κάποια λεγόμενα αποθετήρια ε, δηλαδή αποθεματικά τα οποία έχουν για να μεταφέρουν εκεί ε, τα χρήματα που μπορεί να τους χρειαστούν σε περίπτωση απρόβλεπτου ακραίου κινδύνου για βελτίωση της ρευστότητα, για παράδειγμα. Είναι μια αποταμιευτική αρχή προφύλαξης ουσιαστικά και ανάλογα με τη φορολογική πολιτική που επιτρέπει κάποια τέτοια μέτρα ή τα όρια της ε, κοινή πολιτικής είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τα, τα 39 μέτρα ασφάλισης ουσιαστικά, Δεν έχει να διδαχθεί τόσο πολλά πράγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά δεν υπάρχει υψηλή απορρόφηση στα κράτη-μέλη. Και τα παραδείγματα μας δείχνουν, για παράδειγμα, ότι στην Αυστραλία και ιδίως εσύ ΣΥΠΑ πολύ μεγαλύτερη απορρόφηση. Υψηλά ποσοστά, μέχρι και 80%. Και στην Ιαπωνία είναι σχεδόν υποχρεωτικό αν όχι επίσημα τουλάχιστον ε, όπως λειτουργεί με βασικές καλλιέργειες. Είναι σχεδόν υποχρεωτική συμμετοχή σε τέτοιου είδους ασφαλιστικά σχήματα και υπάρχει και στην αλληλεπίδραση με μέτρα πρόληψης. Οι αγρότες ε, χρειάζεται να κάνουν κάποιες μετρήσεις ε, με υποχρεωτικό τρόπο για τη συγκράτηση του κινδύνου. σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Αυτό που θεωρήσαμε ενδιαφέρον είναι μακροπρόθεσμα. Έχουμε αυτά τα περιβαλλοντικά κλιματικά εργαλεία, έχουμε και τα οικολογικά προγράμματα ετήσιας βάσεις, Το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το αμερικανικό και το αυστραλιανό πρόγραμμα είναι ότι έχουν πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα που κρατάνε 20-30 χρόνια. Για το land consolidation το λεγόμενο. Αν το δούμε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία οικολογικού κεφαλαίου ή την προστασία του κλίματος, Αυτά σίγουρα είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση και χρειάζονται τέτοιου είδους ε, μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, αν μπορώ να τις πω έτσι. Και θα ήταν ίσως ενδιαφέροντα εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε επίσης ε, στον μηχανισμό επιλογής ε, Αυστραλία ή το είπε και Σιμών, έχουν ένα σύστημα πληστηριασμών. Μπορούν δηλαδή να προσφέρουν τις υπηρεσίες του οι αγρότες με κάποια τιμή. σε ό,τι αφορά και εργοπεριβαλλοντικά ε, πράγματα. Όταν έχουμε ένα ειδικό συγκεκριμένο τόπο άσκηση ε, κάποιες δραστηριότητας, ε, μπορεί να μην είναι ίσως το πιο πολλά υποσχόμενο αυτό το μέτρο πληστηριασμών, αλλά όταν θέλουμε να μετριάσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι ένα δημόσιο αγαθό, το που γίνεται συγκεκριμένα, ποιος είναι ο τόπος δεν ενδιαφέρει τόσο. Οπότε εκεί ναι, μας ενδιαφέρει η σχεση κοστος κόστους-οφέλους. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση λοιπόν. Αλλά αυτό ακόμη δεν το έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα, για να το βρω, μείωση κινδύνων ήταν μείωση γεωργικής προέλευσης αέριων και μείωση κινδύνων και στην Ελβετία υπάρχει συνεργασία. Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα, υπάρχουν πιλωτικές προσεγγίσεις για συνδυασμό γνώσης και στήριξης και καινοτομία. Έχουμε κάτι παρόμοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το EIP ε Agri, αλλά έχουμε να διδαχθούμε νομίζω από αυτό το παράδειγμα της Ελβετίας. Ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα είπε η Σιμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καλό επίπεδο βρίσκεται. Όμως και εδώ έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να μάθουμε σε ό,τι αφορά μια συνεργατική δράση και προσέγγιση που βλέπουμε στο Ιαπωνέζικο, για παράδειγμα, πρόγραμμα, όπου τα κονδύλια δεν δίνονται σε μεμονωμένους αγρότες, αλλά ε, σε μια κοινότητα που αναζητεί την καλύτερη δυνατή λύση για μια συγκεκριμένη περιοχή. Βλέπουμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις υπάρχουν διαφοροποίησεις. Δεν λένε δηλαδή πληρώνουμε τους αγρότες ε, για ένα μέσο ε, εισόδημα, αλλά έχουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτερότητες και διαφορές σε ό,τι αφορά τις συνθήκες παραγωγής. Και εδώ νομίζω ότι μπορώ να ολοκληρώσω και να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση και διεξοδική το τέλος, μέχρι τέλος για να έχουμε μία συνολική εικόνα. Ε, όσοι θέλουν μπορούν να παρέμβουν τώρα. Έχουμε 12 ομιλητές, από ό,τι βλέπω στον κατάλογο, Τρία λεπτά για τον καθένα. Παρακαλώ. Για να έχουμε χρόνο και για τις απαντήσεις. Η κυρία Σάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και του ομιλητέ μα εδώ σήμερα το πρωί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό όσα μα είπαν. Για τον τελευταίο καιρό ακούσαμε πάρα πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση τη ε, αγροτική πολιτική στην Ευρώπη. Έχω τρει συγκεκριμένε ερωτήσει ε, προ τον Ρούλ. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση κινδύνου, είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο αυτό το οποίο αναφέρατε και παρουσιάσατε. Θα το εισάγουμε, πρέπει να το εισάγουμε πώς διαχειριζόμαστε τις ε, ε, ομάδες αυτές γεωργών και μιλήσατε και για αποθεματικά. Τι θα κάνουμε στην Ευρώπη. Κατά δεύτερον, το περιβάλλον και το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα της μακροπρόθεσμης αυτής διάστασης στη γεωργική πολιτική σε ό,τι αφορά και τον Γεωργό. Είσαστε από την Ολλανδία. Αν δεν υπάρχει αυτή η μακροπρόθεσμη διάσταση, ουσιαστικά θεωρείτε ότι πρόκειται για δεσπάθηση ε, χρήματο, ότι κατασπαταλάτε τα χρήματα του προλογούμενου. Είσαστε υπέρ. Λοιπόν, τρίτο σημείο τώρα. Στην ε, Βόρειο Ολλανδία συνομιλούμε με μεγάλους ενώσεις γεωργών. Μιλήσατε για εκπομπές, αλλά στην τελική ανάλυση, οι γεωργοί θέλουν να μείνουν γεωργοί. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα εργαλεία που, έχουμε, που παρουσιάσατε για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους παρουσιαστές για αυτή τη μελέτη ακούσαμε από ένα γαλλικό ερευνητικό Ινστιτούτο ε, ότι η Κίνα δαπανά το διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, τομέα της γεωργίας και αυτό ισχύει και για τις ΗΠΑ. Από την δεκαετία του 80 όμως εμείς έχουμε μειώσει την υποστήριξη στην αγροτική οικονομία. Μιλάμε για περικοπές της τάξης του 11% τώρα, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Πώς έχει το συγκριτικό μας πλεονέκτημα υπάρχει καταρχήν. Είμαστε μεταξύ των πρώτων πέντε ή βρισκόμαστε πολύ πιο πίσω. Θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχω ήδη θίξει αρκετές φορές. Μιλήσατε για την Ιαπωνία και για άλλες χώρες και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη γενικότερα ως προς την αγροτική έρευνα. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κλιματικών αλλαγών. Έχουμε μεγάλα προβλήματα ξηρασίας ακόμα και εδώ στην Ευρώπη. Και τώρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται τόσο μεγάλα αρδευτικά έργα. Μιλάμε για ένα μέσο όρο 6,1% άρδευσης. Είμαστε πολύ πιο πίσω από τον μέσο παγκόσμιο όριο. Τι γίνεται ως προς την ποσοστή αναλογία χρήσης αρτευτικών έργων σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και ε, κατά πόσο μπορούμε ε, να έχουμε μέτρα συντήρησης, αποθήκευσης, αποθήκευσης υδάτων. Πώς βρισκόμαστε παγκόσμια. Ευχαριστώ, ο κύριος Μπούντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και εγώ και θα ε, ήθελα να σταθώ και σε ε, ένα θέμα που έθιξε η κυρία Σράιερ, δηλαδή τη διαχείριση κινδύνου. Στον Καναδά μεταφέρεται αυτή η πίεση των χαμηλών τιμών προς τους καταναλωτές. Πότε γίνεται αυτό πόσο χρόνο μάλλον χρειάζεται. Γιατί αν, αυξάνεται η, αν αυξάνονται οι τιμές πέφτουν οι πωλήσει. Άρα ο αγρότης χρειάζεται υποστήριξη σε καθημερινή βάση για την εκμετάλλευσή του, για την εκτροφή των ζώων και ούτω καθεξής. Πώς το θέμα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα. Είπατε ότι οι αγρότες μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν σε καιρό κρίσης. Ποιος τα βάζει τα χρήματα ο αγρότης, ε, γιατί αλλιώς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ο, καθένας, ε, ο κάθε αγρότης μπορεί να βάλει τα χρήματά του στην αποταμίευση. Εμείς πώς συνδράμουμε. Ε, πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχέδιο υποστήριξης των αγροτών. Πώς προωθείται αυτό, πώς ε, ε, υπάρχουν ασφαλιστήρια υπέρ των αγροτών. Τι κάνουν οι ασφαλιστικές ε, εταιρείες, γιατί αυτό το αντιμετωπίζουν Πίσαμε και στην Ρουμανία. Δηλαδή έχουμε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες όπου ασφαλίζονται οι αγρότες και αν δεν έχουν μια ελάχιστη τιμή πώληση, τότε παρεμβαίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Θα ήθελα να μου το διευκρινίζετε αυτό. Σε σχέση με αυτή την αναγέννηση, μάλλον την, τις νέες γενιές που εμπλέκονται στην αγροτική οικονομία, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο υπάρχουν συνεφείς ε, μηχανισμοί, έτσι ώστε να μην έχουμε μέσο όρο ηλικία του αγρότη τα 70 χρόνια όπως ισχύει στην Ιαπωνία, Προσπαθούμε να βρούμε μηχανισμούς για να δελεάσουμε τους νέους στην αγροτική οικονομία, η οποία δεν είναι και τόσο ελκυστική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που είναι ε, ενδιαφέρουσα. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από τις άλλες χώρες ε, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αφήνει την ε, αγροτική οικονομία στους κλειδονισμούς των τιμών. Όλες οι χώρες μετά την κρίση του 7-8 υποστήριξαν τους αγρότες έτσι ώστε να μην υπάρχει κατάρρευση τιμών. Η αγροτική οικονομία πρέπει να υποστηριχθεί. Θεωρείται στρατηγικός τομέας παντού εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ΗΠΑ, Βραζιλία και Κίνα ε, έχουν, έχει αυξηθεί η υποστήριξη από το 2008 και μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μείωση 18% μεταξύ 8 και 15% και αυτή η καθοδική πορεία συνεχίζεται. Η μελέτη που έγινε από το Ινστιτούτο Μοναγκρή δείχνει ότι στις χώρες που προανέφερα θα πρέπει να προσθέσουμε και τη Ρωσία που ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση για το εμπάργο που της έχει επιβληθεί. Επίσης ε, έχει ε, υπάρξει ένα ειδικό νομοθέτημα στις ΗΠΑ υποστήριξης ε, της ε, γεωργικής οικονομίας στο, στη Βραζιλία, Ινδία και ε, Κίνα βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση υποστήριξη και δυστυχώς δεν λαμβάνονται πάντα υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες. Βλέπουμε ότι ότι ο ΠΟΕ ε, λαμβάνει υπόψη την κατάρρευση της παγκόσμιας αγοράς όμως έχουν γίνει πολλές ε, μελέτες υποστήριξης. Εμείς τι περιμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υπάρχουν πια αγρότες για να τους υποστήριξουμε. Thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έγγραφο είναι πολύ χρήσιμο για να μας πείτε τι κάνουν οι διάφορες χώρες για να υποστηρίξουν την γεωργία. Με ενδιαφέρει το θέμα της Αυστραλίας, λέει ο κύριος Άγνιου. Βεβαίως, δεν θα αλλάξουν τον κόσμο και το κλίμα, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο, πώς μάλλον αντιμετωπίζουν τα καύσιμα και τι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να κάνουν για να τύχουν υποστήριξης. Υπάρχει και το θέμα του set aside για να μειωθεί η παραγωγή, δηλαδή να εγκαταλειφθούν οι υγιές για ένα χρονικό διάστημα. Ένας συνάδελφος από τη Ρουμανία μίλησε για τα ύδατα τα οποία δεν υπάρχουν εν αυθονία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε νέο τρόπο παραγωγής καλλιεργειών. Δυστυχώς το πράσινο λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο ισχυρό που έχει καταφέρει να απαγορεύσει τους γενετικούς, τροποποιημένου τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό θα οδηγούσε σε μείωση Χρήση των υδάτων. Δεν θα πρέπει να κατασπαταλούμε τα χρήματα εκεί που μπορούμε να αποταμιεύσουμε. Αν δείτε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βραζιλία θα μπορούσε να υποστηρίξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή υπάρχει η ε, αμυψισπορά, και τα σχέδια υποστήριξης και αποταμίευσης. Όμως υπάρχει και, το, και η άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή ε, οι κλιματικές αλλαγές και βεβαίως ε, η διατροφή και τα τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Δηλαδή κάποια στιγμή η Βραζιλία να προτάσει και να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται διατροφική ασφάλεια για πολλές χώρες. Αυτό θα ήθελα να αναφερθεί. Πάντα ε, υπάρχουν αντισταθμίσματα. Θα πρέπει να υπάρχει διατροφική ασφάλεια από όλες τις ε, χώρες, αλλά τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν λογικές τιμές. Θα πρέπει να φύγω για λίγο, αλλά θα έρθω για να ακούσω τις απαντήσεις. Κολομπιέ. Ναι. Σε αυτή την έκθεση, κύριε Πρόεδρε, διάφορες σταθερές βλέπουμε για τη γεωργία που τα πάνε πολύ καλύτερα ε, τα πράγματα άλλες χώρες από ότι εδώ, στήριξη της τιμής αγοράς, το αντίθετο στη χώρα στο ΩΣΑ, αλλά ο μηχανισμός αυτός προστατεύει τους γεωργούς ε, και τα εισοδήματά τους. Οι συστάσεις της μελέτης τρία βασικά σημεία αναφέρουν τα σχέδια κάλυψης κινδύνων, τα, σχέδια, τα εργαλεία διαχείρισης ατομικοικών αρχείων άνθρακα και αποζημιώσεις για φυσικές ελλείψεις. Όμως αυτό αρκεί πάντα με οπτική την μελλοντική ΚΑΠ για τον καθορισμό μιας πραγματικής γεωργικής πολιτικής. Δεν νομίζω. Τι γίνεται με τη ρυθμίση των αγορών και πώς επηρεάζουν τα έσοδά τους. Τα είπα. Τι κάνουμε με την ποιότητα των τροφίμων την ανανέωση τη δεγενειακή στη Γεωργία. Τίποτα. Και πιο πολύ γίνεται λόγος για ιδιοκτήτες γεών στην έκθεση και όχι για αγρότες. Ενώ η παραγωγή τροφίμων φαίνεται κάτι δευτερεύον για τους ε, συντάκτες της έκθεσης. Άλλη πτυχή των εξελίξεων. Ότι όλες αυτές είναι συμβατές με τον ε, άκρατο φιλελευθερισμό που δεσπόζει στην Ευρώπη και την ε, άναρχη επίσης ε, ε, υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση. Εγώ νομίζω ότι η γεωργία και η υπεθρός πεθαίνουν και αυτή είναι πραγματικότητα γιατί λείπουν πολιτικές που εδράζονται στην γεωργική παραγωγή. Δική μας ευθύνη των πολιτικών είναι να εστιάσουμε την πολιτική στους ενεργοί αγρότες και στην παραγωγή τους. Έχουμε πολλά παραδείγματα καλά. Αν δεν γίνουν αυτά, θα ε, γυρίζουμε άσκοπα ε, σε φαυλοκύκλο. Και οι πολύ μεγάλοι γεωκτήμονες ε, θα συγκεντρώνουν γέες για να πλουτίζουν με επιδοτήσεις σε βάρος των τοπικών κοινωνιών και σε βάρος της οικογενειακής γεωργίας που στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ε, είναι η πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ε, Κύριος Φλάναγκαν, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και πολύ καλή. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων και τα σχετικά εργαλεία, έχουμε πολλές αναφορές σε χρηματοδοτικά εργαλεία και στις νέες προτάσεις ε, της κοινής γεωργικής πολιτικής. Πριν ακολουθήσει κανείς αυτό το μονοπάτι κοιτάζει, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος θέλει να μετακινήσει μια καρότσα, δεν ψάχνει ε, ένα τετράγωνο, ψάχνει ένα τροχό, που είναι ήδη κάτι που έχει εφευρεθεί. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν δουλεύουν πολύ καλά. Ε, στον Καναδά και στη ΣΥΠΑ έχουμε εργαλεία ε, διαχείρισης κινδύνων. Πώς βοήθησε αυτό τους γεωργούς στις χώρες αυτές. Ε, το έχω πει και στην Κομισιόν. Τέτοια πράγματα θα δούμε και εδώ, σαν αυτά που βλέπουμε στην Αμερική. Έχουμε τον Tiger Woods και τον Rory McIlroy και άλλους που παίρνουν χρήματα από τη γεωργική ασφάλιση ε, και έχουν κάποια κονδύλια των 2 εκατομμυρίων που τους διατίθενται. Πού τα βρήκανε, τι ε, πρόθεση έχει η Κομισιόν να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και γιατί. Και βλέποντας τι γίνεται στον κόσμο και τι γίνεται στην Ευρώπη, έχουν οι ομιλητές κάποια παραδείγματα για προγράμματα στήριξης που πληρώνουν τον κόσμο για το τι έκανε πριν 20 χρόνια. Γιατί αυτά κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε, υποτίθεται, με την αλλαγή της ΚΑΠ ε, και θα αλλάξουν πολλά. Αλλά διπλή γλώσσα, διγλωσία ε, βλέπω όλοι είναι κατά του να, να πληρώσουν τους αγρότες για αυτά που έκανε το 2001 ή το 2002. Αλλά δεν θέλει κανείς να το αποτρέψει για το μέλλον και μάλλον θα γίνει με αυτά τα οικολογικά σχέδια. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μοντέλο στον κόσμο. Πληρώνει, υπάρχει άλλο μοντέλο που πληρώνει τον κόσμο για το τι έκανε πριν 20 χρόνια και όχι το τι κάνει τώρα. Ένα άλλο ενδιαφέρον της παρουσίασης ήταν αυτό το σχέδιο παγίδευσης άνθρακα στην Αυστραλία. Έχετε ε, κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Δύσκολα θα περιληφθεί στη νέα κάποια την αργά. Θα έπρεπε όμως, γιατί στην Ιρλανδία ε, και φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές της και σε άλλα μέρη του κόσμου το ίδιο συμβαίνει. Δίνονται κίνητρα στον κόσμο για να παράγονται, μάλλον για να καλλιεργούνται κάποια ε, φυτά που παράγουν 12.000 ε, τόνους οξυδίου ε, του άνθρακα, ενώ υπάρχουν 40.000 τόνοι άνθρακα που παγιδεύονται ήδη εκεί. Άρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι θετικό. Θα έπρεπε να έχουμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και είναι κρίμα πραγματικά που ο συνάδελφος Αγνιού έφυγε. Ίσως να πήγε στο γραφείο του για να κάνει τα μαθήματά του. Δεν υπάρχει απαγόρευση των γαματάφα κατά όμικρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μόνο ένα θέμα πρόληψης κινδύνου. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όμως ό,τι αφορά την ασφάλεια σε τεφαρά τους κινδύνους. Υπάρχει ένα ποσοστό των πόσων χρηματοδότησης που φτάνει στους αγρότες. Τι πόσο δηλαδή καταλήγεται στους αγρότες και τι πόσο απορροφάται από τις ιδιωτικές ε, εταιρείε. Και δεύτερον, έχετε συγκρίνει άλλα μέτρα και άλλες στρατηγικές για την παροχή χρημάτων στους αγρότες σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ των στόχων της, ε, του περιβάλλοντος και τον στόχο του να μείνουν οι αγρότες ε, στην Ήπεθρο. Έχετε λοιπόν κάποιο δίκτυο για το τι είναι πιο επιτυχές ε, ως μέτρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελαή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους δύο πανελίστες για την παρουσίασή τους. Αμφιβάλλω ωστόσο πρέπει να πω. Μας μιλάτε για εργαλεία. Για την αρχή της πρόληψης, η τελική ανάλυση. Δεν μας ε, μιλάτε όμως για τη σύγκριση των χρηματικών πόρων στις χώρες που εξετάσατε. Και αυτό προφανώς έχει μεγάλες αντικτύπω σε ό,τι αφορά τη χρήση, την αξιοποίηση των εργαλείων για τη διαχείριση του κινδύνου και για την πρόληψη. Και όλη αυτή η παρουσίαση με οδηγεί σε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Οι χώρες αυτές ε, που εξετάστηκαν, τι έχουν ως πραγματικό απότερο στόχο. Είναι η ανεξαρτησία σε επίπεδο τροφίμων, ε, η σχετική πολιτική για την γεωργία και για τα τρόφιμα, για να υπάρχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Εκεί μιλάμε πιο πολύ όχι τόσο για γεωργική πολιτική, αλλά για περιβαλλοντική πολιτική. Άρα είναι δύσκολο να επιδιώξουμε όλους τους στόχους ταυτόχρονα με το ίδιο επίπεδο δέσμευσή. Και εγώ θα ήθελα στην Ευρώπη να ξέρουμε τουλάχιστον πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Και να χρησιμοποιήσουμε τελικά τους ε, δημόσιους πόρους για να δημιουργήσουμε ε, ένα δίκτυο γεωργικό γιατί μας ταιριάζει, γιατί μας δίνει ένα καλό επίπεδο τροφίμων, μια αυτονομία σε επιστηστικό επίπεδο. Αυτό αποτελεί διαφορετικό στόχο προφανώς. Καταλαβαίνω τι μας λέτε και τα πορίσματα τα οποία εξαγάγανται, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουμε πρέπει εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τι θέλουμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά τη Γεωργία. Ντόκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. αυτή μας δίνει, η, η μελέτη μας δίνει μια καλή εντύπωση για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτό που λείπει ωστόσο είναι η Λατινική Αμερική, η Νότιος Αμερική, που έχει μεγάλο αντικτύπο προφανώς ε, στο τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά η συμφωνία Μερκοσούρ που επίσης ε, μπορεί να έχει γενικότερε επιπτώσεις. Πείτε μας δύο λόγια. Κατά δεύτερον, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τη σχέση μεταξύ των διαφορών σχεδίων ε, υποστήριξη και τη γεωργία. Ω τώρα δεν είχαμε στην Ευρώπη ένα σύστημα που να βασίζεται στην παραγωγή ο δεύτερος πυλώνας είναι η ανάπτυξη τη υπέτρου και το τρίτο σκέλο ο τρίτος πυλώνας, όλο και πιο πολύ έχει να κάνει με το περιβάλλον. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς δημιουργούνται οι ισορροπίε μεταξύ των τριών αυτών σκελών στις χώρε που εξετάσατε. Άρα άμεσε πληρωμέ ε, στου γεωργού Δεύτερον, το περιβάλλον και η ανάπτυξη τη υπέτρου. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα με ενδιαφέρει είναι η γραφειοκρατία που ενέχεται στα συστήματα αυτά. Εκ πρώτης όψεως, τα συστήματα αυτά που αναλύσατε φαίνεται ότι είναι κάπως πιο απλά. Και γνωρίζουμε από τις συνομιλίες μας με τους αγρότες ότι το πρώτο πράγμα το οποίο καταγγέλουν είναι ότι η ΚΑΠ είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γραφειοκρατία από αυτό που θα θέλαμε. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε τι γραφειοκρατία χρειάζονται, τι ποσοστό γραφειοκρατία αντιμετωπίζουν συγγνώμη, οι άλλε χώρε. Ε, φυσικά ε, επιμένοντα στο σκέλο τη απλοποίηση. Και ύστερα, όπω ε, υπογραμμίσατε και εσεί στα συμπεράσματά σα, όλα τα συστήματα τα οποία μελετήσατε έχουν ε, κάποια μορφή ασφάλειας ε, από κινδύνου, είτε κινδύνου τη αγορά, είτε κινδύνου από φυσικέ καταστροφέ. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε εμεί στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Και διαπιστώνοντα ότι όλο και πιο πολλά όλο και πιο πολλοί πόροι αφιερώνονται στην ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Δεν συμφωνείτε ότι κάποια συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτές τις πιο πλούσιες χώρες είναι πολύ πιο γενναιόδωρα στη τελική ανάλυση από τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα συστήματα. Ο κ. Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ήθελα να ευχαριστήσω και τους προσκαλεσμένους μας ε, για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τις συστάσεις τους. Μιλάμε ε, για διαχείριση κινδύνου και εποπτεία κινδύνου. Δυστυχώς αυτό είναι πολύ περιορισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ε, λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφαρμογή αυτών των ε, μέτρων με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να συζητηθούν σε εύρος αυτά τα ζητήματα. Διαφορετικά δεν θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Και έχω και μία ερώτηση σε σχέση με την υποστήριξη ε, αγροτικών κοινοτήτων. έγιναν επιπρόσθετες ε, καταβολές εκεί που χρειάζεται, εκεί που χρειάστηκε και τι καταβολές έγιναν, τι πληρωμές έγιναν ξεχωριστά εκεί που χρειαζόταν στους γεωργούς μέσα στα πλαίσια των σχεδίων υποστήριξης. Επίσης προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε μέτρα διαχείρισης κινδύνου στον γαλακτοκομικό τομέα κάτι το οποίο λειτουργήσε πολύ καλά. Θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε μαθήματα από αυτή την εμπειρία μας. Στη χώρα μου και στις βόρειες και ανατολικές χώρες έχει μεγάλη ε, σημασία η παροχή τροφίμων που να σχετίζεται και με το γεωργικό τομέα αλλά και με τον τομέα της εκτροφής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι τι έχουμε, τι υπάρχει στην Αυστραλία ή στην Ελβετία, αλλά τι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς διαθέτουμε την ΚΑΠ αλλά τα σχήματα υποστήριξης είναι διαφορετικά. Αλλάζει και η τάξη μεγέθους των συστημάτων άμεσων πληρωμών στα κράτη-μέλη, γιατί πολλές φορές χρειάζεται υποστήριξη δυνάμει του δεύτερου πυλώνα και άλλα κράτη-μέλη προσπαθούν να ε, συμπληρώσουν αυτό το σχήμα μέσω των γεωργικών υποδομών. Άρα θα ήταν ίσως καλύτερα αν θα μπορούσε να συγκρίνει την κατάσταση κανείς στις πέντε χώρες που εξετάσατε με την κατάσταση ε, σε άλλα κρατή-μέλη, δηλαδή πώς η Αυστραλία μπορεί να συγκριθεί με την Πολωνία ή την Ισπανία. Έτσι η σύγκριση θα γινόταν πιο εύκολη, γιατί η ΚΑΠ αφήνει πολλά περιθώρια στα κράτη-μέλη, υπάρχει διακριτική ευχέρεια, ιδιαίτερα στις πλέον απομακρυσμένες ε, περιοχές. Άρα η κατάσταση στα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς. Και ποιος παίρνει αυτή την υποστήριξη, οι αγρότες ή οι ιδιοκτήτες, ε, οι γεωκτήτες. Στο άρθρο 16 της Συνθήκης Προσχώρησης αναγράφεται ότι δίνεται ενίσχυση στους εργαζόμενους ε, κάθε αυτούς. Αν λοιπόν ο αγρότης προσλάβει κάποιον ε, για ε, την γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων είναι, θα μπορούσε να είναι επιλέξιμος ή όχι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ήμουνα σε όλη την παρουσίαση αλλά με βάση αυτά που συζητάμε και σε συνέχεια αυτών θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια και να υποβάλω ερωτήσεις. Ενώ η αγροτική ε, στην ουσία η οικονομία και πολιτική δίνει ενισχύσεις και μόνον δεν επιλύουμε το θέμα. γιατί Χρειάζεται να δούμε την κατανομή αυτών των ενισχύσεων. Πολλές φορές είναι άδικες, όμως το δημόσιο χρήμα που χορηγείται στους αγρότες στην ουσία δεν είναι για αυτούς, αλλά για να έχουμε φτηνή πρώτη ύλη στα χέρια μιας βιομηχανίας η οποία θα βοηθήσει τη μεγάλη βιομηχανία εξαγωγών. Αυτό θα πρέπει να το πούμε σαφώς, γιατί εμείς λέμε στους αγρότες, ε, κυρίες, κύριοι, ε, δουλεύετε δωρεάν σχεδόν, γιατί οι τιμές των προϊόντων σας είναι σχεδόν μηδενικές. Θα εργαστείτε δωρεάν. Αυτό τους λέμε. Και μετά θα δούμε κατά πόσο υπάρχει δημόσιο χρήμα για να αντισταθμίσουμε αυτό, το, αυτή, τη, αυτή την δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Άρα, αυτό έχει ε, επιπτώσεις, ε, μιλάμε για απερίμωση, για αύξηση της μέσης ηλικίας των αγροτών. Ποιους ε, τεχνικούς λόγους μπορείτε να προβάλλετε για να μην μιλάμε για τιμές που καλύπτουν το κόστος της παραγωγής, γιατί η κοινωνία πληρώνει διπλά. Πληρώνει τα τρόφιμα και πληρώνει με μία φορολογία αυτή την βιομηχανία που έχει φθηνή πρώτη ύλη. Θα πρέπει να το πούμε αυτό σαφώς, διότι έχουμε βαρεθεί να ακούμε τα ίδια. Θέλω να μου εξηγήσετε ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το θέμα έτσι ώστε να μην έχουμε τιμές ε, που να χορηγούν αντισταθμίσματα. Θα πρέπει να δούμε ποια πολιτική θέλουμε, να το αποφασίσουμε αυτό. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, λέει ο πρόεδρος, σε αυτή την περίπτωση θα παρακαλέσω τους δύο ομιλητές μας να απαντήσουν ε, στις ερωτήσεις, στα σχόλια και να κάνω και κάποια σχόλια για τη μελλοντική κυνηγιορική πολιτική. Βέβαια όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εμείς ε, γιατί καταθέτουμε και τροπολογίες ε, και σύντομα θα ψηφίσουμε κιόλας ε, για την κοινή γεωρική πολιτική. Και η εμπορική συμφωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο, όπως και η φορολογία, θα επηρεάσει σημαντικά. Και η γεωργία στις διάφορες χώρες. Αυτά από πλευρά μου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας αυτές και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου και τη διαχείριση των οικονομικών. Ένα σχόλιο της κυρίας Σχράιερ για τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Αυτά νομίζω θα τα επεξεργαστή συνάδελφο. Αλλά σίγουρα αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθεί όμως αυτό ως ε, πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά και το συνδυασμό με το Natura 2000 και σε ό,τι αφορά τα τρυφόδια εδάφη. Σε ό,τι αφορά και τι μακροπρόθεσμε δεσμεύσει, αυτό φυσικά επηρεάζει. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την διαχείριση κινδύνου, γιατί ετέθησαν πολλές ερωτήσεις ε, στο σημείο αυτό. Ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό ενδεχομένω θα πρέπει να το κάνουμε πιο πολύ και σίγουρα γίνεται αυτό στη ΣΥΠΑ, το έθεσε και ο κ. Φλάναγκαν στην ερώτησή του. Τι συνολικός όγκος χρημάτων τελικά καταλήγουν στις ασφαλιστικές. Δεν έχω ακριβή αριθμητικά στοιχεία υπόψη μου. Κάναμε μια σχετική μελέτη πρόσφατα για την Γενική Διεύθυνση Άγκρη και έχει να κάνει με το θέμα αυτό. Αλλά είναι ψηλό το πόσο και όντω θα πρέπει να κοιτάξουμε το κόστο συναλλαγή. Είναι πολύ ψηλό σε κάποιε περιπτώσει. Και φυσικά είναι και το θέμα του κατά πόσο υπάρχει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα για το πρόγραμμα. Χρησιμοποιούν λοιπόν και δημιουργούν μεγαλύτερο, μεγαλύτερη απορρόφηση στην Ευρώπη. Αλλά στην τελική ανάλυση αξίζει τον κόπο. Εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν ε, τι γίνεται. Γιατί πραγματικά υπάρχουν λόγια ανησυχία για το σύστημα του, τον ΙΠΑ. Άλλο ένα σχόλιο το οποίο ακούσαμε. Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικό σύστημα γιατί με τις άμεσες πληρωμές ήδη ενισχύουμε τους αγρότες. Εδώ θα ήμουν πιο επιφυλακτικός. Και αυτό γιατί εγώ πιστεύω ότι η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να οδηγεί σε, διαχείριση, σε ασφάλεια σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος. Και ασφάλεια, ας πούμε, θα ήταν ένα σύστημα αμα, για τη διαχείριση κινδύνου. Αλλά αυτό που κάνουν ε, προφανώς είναι ότι συμπληρώνουν και το εισόδημα των γεωργών. Σταθεροποιούν το εισόδημα των γεωργών. Αλλά οι άμεσες πληρωμέ προφανώς έχουν και άλλους στόχους. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν δεν θα πρέπει να προκαλείται σύγχυση με τα μέτρα αυτά. Έγιναν και κάποιες ερωτήσεις ε, για το σύγκριση που έγινε γιατί τα κατά πόσο μπορούν να μεταφερθούν τα απορίσματα από πανδημία, έρευνα και να χρησιμοποιηθούν στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη φυσικά η κατάσταση είναι πολύ ιδιαίτερη. Φυσικά αυτό ισχύει. Και γι' αυτό λοιπόν στην Ευρώπη, στην μελέτη μας, χρησιμοποιήσαμε και την προσέγγιση με τον πίνακα για την διαχείριση κινδύνου, για παράδειγμα. Κοιτάμε διάφορες χώρες αν θέλουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο για τον αγρότη, τι είδου μέτρα χρησιμοποιούν. Και μετά προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σύγκριση. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορέ. Αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ήταν χρήσιμο να υπάρχει ε, αυτό το εργαλείο, αυτός ο πίνακα σύγκριση ε, μέτρων ανάλογα με το στόχο. Ένα από τα στοιχεία που ακούσαμε ήταν για την ε, οικονομική πολιτική Είπε κάποιο ότι δεν θα έπρεπε μήπως να κοιτάξουν πιο πολύ την οικονομική πολιτική, γιατί υπάρχει φυσικά διαπαφή μεταξύ τη οικονομική ε, πολιτική και τη διαχείριση κινδύνου. Ναι. Κοιτάμε και πέρα από τη γερική πολιτική. Κοιτάξαμε και πέρα από τη γερική πολιτική στην ε, έρευνα μα, όχι μόνο για τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά για τι επενδύσει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε γιατί σε κάποιε χώρε οι γεωργοί επενδύουν πιο πολύ σε σχέση με άλλε χώρε. Νομίζω ότι τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κινητήρα και για τις επενδύσεις και για το λόγο αυτό και για την καινοτομία κατά συνέπεια στον τομέα των, της γεωργίας. Υπάρχει, για παράδειγμα, και χώρες που χρησιμοποιούν φορολογικά κίνητρα. Νομίζω λοιπόν ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε καλύτερα για να έχουμε επίσης και επίγνωση του τι ήδη υφίσταται, τι ποια μέτρα υφίσταται και ποιος είναι, ποια είναι η σχέση με τα δικά μας μέτρα. Γιατί μπορεί σε τελική ανάλυση να υπάρχουν κάποιες διαφορές στην αντιμετώπιση των γεωργών. Υπάρχει και το θέμα φυσικά των ίσων όρων ανταγωνισμού. Φαντάζομαι ότι αυτό σας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο. Κάποιο σχολίασε το, το γεγονός ότι δεν κάναμε πιο πολύ έρευνα στην Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά εφαρμογή τη έρευνα. Είχαμε περιορισμού. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχουμε εξετάσει πιο πολύ και το σκέλο αυτό. Και τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο. Μάλιστα. Εγώ θα προσπαθήσω να ακολουθήσω λίγο τα ίδια αυτά επιχειρήματα των ήρμων των σκέψεων του προαλήσαντα συναδέλφου μου για τους ε, στόχους της πολιτικής για την ισορροπία, το θέμα της ασφάλειας τροφίμων ε, και τους στόχους εκεί έγιναν κάποια σχετικά σχόλια. Στην παρουσίαση ήδη είπαμε πως ξεκινήσαμε από τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτή ήταν η αφετηρία μας για να δούμε τι εργαλεία έχουν οι διάφορες χώρες σε σχέση με αυτό. Είδαμε όμως και τη διαφορά των στόχων της ΚΑΠΑ στις χώρες. Βέβαια, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Στην Αυστραλία, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, έχουν ένα πολύ ισχυρό οικονομικό στόχο και Ελάχιστες είναι οι περιβαλλοντικές πτυχές της γεωργικής πολιτικής, γιατί είναι εκτός πεδίου γεωργικής πολιτικής περιβαλλοντική στόχη. Στον Καναδά συνδυάζουν τους οικονομικούς στόχους με λίγους ε, περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς στόχους, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη έμφαση όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Παπονία και η Ελβετία μάλλον μοιάζουν περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συνδυάζουν ε, τις δύο δέσμες στόχων. Και για τη ΣΥΠΑ το ενδιαφέρον είναι ότι εστιάζουν ιδιαίτερα στην ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο των γεωργικών στόχων. Αυτό δεν είναι τόσο προεξέχον στις άλλες χώρες. Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η Ελβετία έχει πολύ μεγάλη έμφαση στους στόχους που άπτονται της προστασίας του καταναλωτή. Ένα είναι λοιπόν οι στόχοι και άλλο είναι τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων. Και δεν υπάρχει ένα έτσι αρμονικό πάντρεμα πάντα. Και ενδεχομένως να υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να διαμορφώνονται ή να αναφέρονται ως στόχοι πολιτικής, αλλά μέσα δεν βρήκαμε, εργαλεία δεν βρήκαμε. Ίσως δηλαδή μια χώρα να λέει ότι είναι πολύ σημαντικός στόχος η ασφάλεια των τροφίμων, αλλά να είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα εργαλεία προς την πρόθεση του στόχου αυτού. Και δεν ε, είχαμε ως στόχο μας να δούμε αν υπάρχει συνέπεια μεταξύ των στόχων και των τρόπων με τον οποίο διώκεται η εφαρμογή τους, αλλά εστιάσαμε κυρίως ε, στο να δώσουμε παραδείγματα από άλλες χώρες, από τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα και για να επανέλθω στην ασφάλεια των τροφίμων στις Ηνωμένε Πολιτείε. αυτό το οποίο είδαμε είναι πως ένα μέρος της γεωργικής πολιτικής έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση και προστασία, παροχή τροφή, σε άπορους, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συμπεριλάβει στην Ένωση εμείς στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής. Ελπίζω ότι απάντησα για τη σχέση μεταξύ των στόχων πολιτικής και της χώρας. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο για την, Κινέζ... για την καναδική γεωργική πολιτική είναι ότι εστιάζει ιδιαίτερα στην απλούστευση, δηλαδή ελαχιστοποίηση των προσπαθειών ε, του οικονομικών ε, για τη σχετική πολιτική. Βέβαια δεν είχαμε ούτε το χρόνο ούτε τα μέσα για να δούμε αναλυτικά τι γραφειοκρατικές προσπάθειες πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή των διαφόρων ε, μέσω την εκτέλεση των διαφόρων εργαλείων. Δεν μπορώ να πω πολλά για την γραφειοκρατία επομένω. Μόνο αν γινόταν ιδιαίτερη μνήμα το είδαμε το θέμα αυτό. Διαβάζω λίγο τις σημειώσεις μου. έγιναν κάποιες ερωτήσεις για κάποια κοινοτικά προγράμματα. Τα είδαμε και αυτά. Δύο τον αριθμό ε, βρήκαμε στην Ιαπωνία και τα δύο, αν δεν απατώμε. Είναι κάτι ενδιαφέρον, μπορούμε να το δούμε και αυτό. Και υπήρχε και ένα άλλο πρόγραμμα. Πρέπει να δω πώς λεγόταν. Για τους καλλιεργητές ρυζιού στην Ιαπωνία. Για τη ένα mutual insurance scheme όπως λεγόταν, αντασφάλιση και ασφάλιση είναι πράγματα τα οποία ε, λαμβάνονται εκεί υπόψη. Ξέρω ότι και στην Ολλανδία, ε, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής, ε, γίνονται ορισμένα πράγματα, θα μπορούσαμε να τα αντιγράψουμε σε άλλους τομείς πολιτικής ανανέωση των γενών υπάρχουν στην Ιππονία κάποια σχετικά προγράμματα, ιδίω για να προσελκυθούν νέοι αγρότες Βέβαια εκεί υπάρχει και η είσοδος της βιομηχανίας ε, και των μεγάλων επιχειρήσεων στη Γεωργία για την πρόθεση της ε, γενναίκης αλλαγής και προωθούνται οι μεγάλες κλίμακας γεωργικές επιχειρήσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γενναίκης ε, αλλαγής ανανέωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να προσθέσω για να δω τι λέω, δω σημειώσει μου. Να προσθέσω εγώ κάτι. Υπήρξε μία ερώτηση. Γιατί υποστηρίζουμε τους αγρότες με βάση αυτά που έκαναν 20 χρόνια πριν. Και γιατί δεν υπάρχει νέα προσέγγιση. Εγώ είμαι οικονομολόγος και από οικονομικής πλευράς κατανοώ αυτή την ερώτηση. Αλλά ένας από τους λόγους είναι ο εξής, δηλαδή το δημόσιο χρήμα πάει για δημόσια αγαθά. Και στο παρελθόν είχαμε αυτό το θέμα του, του υποδείγματος ε, εσόδων με βάση δηλαδή την παραγωγικότητα και τη στιγμή που υπήρχε αύξηση παραγωγής. Ήμασταν πολύ, είχαμε μεγάλη επιτυχία με αυτή την αλλαγή και τώρα ε, δεν ε, έχουμε σταθεί σε αυτό το παράδειγμα εσόδων. Θα πρέπει να δούμε τους αγρότες πιο θετικά, όχι ότι είναι ε, θύματα και στο Ταμείο Ανεργίας παρέχουν οι υπηρεσίες, αυτό είναι θετικό, και στους δώσουμε κίνητρα με βάση αυτό που κάνουν. Εάν παρέχει κανείς, ε, ε, αν παρέχει αυτά τα δημόσια αγαθά, θα πρέπει να ανταμείβεται. Και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουμε και στα πλαίσια της επανακατανομής. Εκεί δηλαδή που παρέχονται υπηρεσίες, ας πούμε στη Ρουμανία, για παράδειγμα, αν μιλάμε για αυτές τις πράσινες υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά, έχετε πολλές περιοχές ε, ποιοτικά πολύ καλές. Θα πρέπει όμως να τις διατηρήσουμε. Στην Ολλανδία διαφορετικά προβλήματα αντιμετωπίζουν, αλλά έτσι θα πρέπει ε, να συνδέουμε το χρήμα. Υπάρχει το θέμα της ε, τιμολόγησης, της πραγματικής τιμολόγησης με βάση την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε συστήματα πληρωμών που να δίνουν ε, κίνητρα στους αγρότες για να αναπτύξουν περισσότερο και καλύτερα την παραγωγή τους. Αυτά. Και Τέλος, υπήρξε μία ερώτηση για αυτά τα χρήματα που μένουν. Τα χρήματα αυτά ε, παραμένουν στη διάθεση του αγρότη, δηλαδή είναι ένας λογαριασμός που διαθέτουν οι αγρότες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα υπό συνθήκες. Αυτό είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως και σε σχέση με την ε, ε, διαχείριση κινδύνων, ίσως ε, στον Καναδά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα με αυτή την καταβολή χρημάτων. Υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει ένα θέμα και θα πρέπει να αποτιμηθεί. Άρα την πληρωμή την παίρνει ο αγρότης ένα-ενάμιση χρόνο μετά. Αυτό δεν βοηθάει τότε τον αγρότη. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ταμιευτήρια, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου που χρησιμοποιείται από τους αγρότες όταν χρειάζεται. Κάτι άλλο που θέλω εγώ να απαντήσω αφορά τις δημοπρασίες στην Αυστραλία για την ανάκτηση ή κατάσχεση άνθρακα. Αυτό αυτό δεν είναι μέρος της ε, αγροτικής πολιτικής, αλλά της πολιτικής αντιμετώπισης του κλίματος. Και τη στιγμή που υπάρχει κατάσχεση άνθρακα, οποιοδήποτε πρόγραμμα, έχει ένα αντίτιμο, δηλαδή μπορεί να απομακρυνθεί μία μονάδα εκτροφής, να γίνει αναδάσωση και ούτω καθεξής. Ε, σε αυτή την περίπτωση δεν διατηρείται η αγροτική παραγωγή, αλλά βεβαίως στην Αυστραλία υπάρχουν ε, τεράστιες εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτατικά και όχι εντατικά. Και αυτό μπορεί να αφορά ε, μία διαδικασία αναδάσωσης Τώρα, ποιος ε, πληρώνει οι γεωκτήμονες ή αυτός που εκμεταλλεύεται τη γη. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε καθε αυτό. Εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε το αντίτυπο στους αγρότες, ανεξάρτητα από το ποιο μέσο χρησιμοποιούν. και ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Άγνιου, κάτι είχε πει και ίσως κάτι θέλει να προσθέσει. Και εγώ έχω μία ερώτηση που ξέχασα να αναφέρω. Ως προς την επιλογή της χώρας, γιατί έχετε επιλέξει μία χώρα και όχι μία άλλη πώς, τι, τι κριτήρια ακολουθείτε, πώς έχει αυτή η διαδικασία επιλογής. Επίσης, οι πληρωμές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους αγρότες, πώς βλέπετε σε σχέση με τον ε, περιβάλλοντα χώρο, πώς ε, μπορούν να γίνουν αυτές οι καταβολές. Ε, Σράιερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω να κάνω ακόμα. Μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. πω θα διατηρήσουμε την επιστημονική ασφάλεια στο άρθρο 2 τη Κλιματική Συμφωνία στην Ευρώπη και ε, διατηρούμε και τι ε, των αγροτών. Αυτό είναι που μας απασχολεί και γιατί το ρωτώ αυτό πριν από κάποιες εβδομάδες ε, στο Παρίσι άκουσα μεγάλες πολυεθνικές ε, που έχουν να κάνουν με την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη και εκφράζουν ε, ε, ότι είναι τόσο υψηλέ οι προδιαγραφέ ε, στην Ευρώπη που θα σταματήσουν σιγά σιγά την παραγωγή. Θα πάνε στην Αμερική, στη Ρωσία, στην ε, Λατινική Αμερική. Και τι θα γίνει τότε, θα μείνει άδεια η υπεθρό μα. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν. Και μήπω έχετε κάνει να προσθέσετε προ την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Ε, αν θέλετε να απαντήσετε στι ερωτήσει αυτέ. Yeah, Ρωτήσατε το θέμα των πληρωμών για τις υπηρεσίες στην Ήπεθρο. Πρέπει να σας πω ότι δεν βρήκαμε πολλά εργαλεία για ανάπτυξη της Ήπεθρου. Όπως την ε, εννοούμε στην Ευρώπη, δεν είναι στο επίκεντρο των γεωργικών πολιτικών στις χώρες. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η έννοια τη ανάπτυξη τη υπαίθρου εξαρτάται πάρα πολύ από την κατανόηση του τι αποτελεί ανάπτυξη τη υπαίθρου. Για παράδειγμα, στην ανάπτυξη τη υπαίθρου στην Ιαπωνία σημαίνει πιο πολύ η ανάπτυξη τη γεωργία. Έχει πολύ έντονα στοιχεία υποστήριξη τη γεωργία. ενώ για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Έχει να κάνει πιο πολύ με επενδύσεις σε επιχειρήσει σε υποδομές και το καθεξής δεν βρήκαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον από πλευρά τη υποστήριξη των ε, περιοχών της υπαίθρου σε ό,τι αφορά τις βασικές ε, υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία στο ιαπωνικό πρόγραμμα. Υπάρχει η πληρωμή πολυλειτουργικότητας και υπάρχει και μια πληρωμή για την βελτίωση την, ε, του εδάφους, αλλά και πάλι με επικέντρωση στη Γεωργία. Αυτό προφανώς και επηρεάζει και την ε, γενικότερη περιοχή της υπέθρου, αλλά δεν έχει τόσο πολύ τη διάσταση τη ανάπτυξη της υπαίθρου. Για το άλλο ερώτημα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τι περιβαλλοντικές δράσεις. Όλες αυτές τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, όλα αυτά τα μέτρα έχουν ως αντίκτυπο προφανώς την αύξηση του κόστους ε, για τους αγρότες και τις ε, παραγωγής ε, τροφίμων. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η γεωργία από πλευρά των εσόδων έχει λίγο πολύ τα ίδια όσο και οι άλλοι τομείς. Αν αυξηθεί το κόστος αλλά όχι το εισόδημα, προφανώς δημιουργούνται εντάσεις και συμφωνώ που επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ενδεχομένω το τρόφιμα είναι πάρα πολύ φτηνά και θα πρέπει να κάνουμε μια εκ νέου αξιολόγηση των τροφίμων προκειμένου να συμπεριληφθεί όλο αυτό το κόστος το οποίο κρύβεται, το οποίο θεωρούμε σημαντικό. Γι' αυτό και έκανα αυτή την ε, σύνδεση, γιατί το θέμα είναι στη τελική ανάλυση ποια είναι η πραγματική τιμή του φαγητού των τροφίμων. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρκετά καλό σύστημα τώρα σε ό,τι αφορά και τους δείχτες που έχουμε στη διάθεσή μας και θεωρώ ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα η ρύθμισή μας στην ε, Ολλανδία, για παράδειγμα. Έχουμε πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής και δείκτες σε ό,τι αφορά την παραγωγή αυτή. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Φρίσλαντ υπάρχει παραγωγή γραφειοκομικών που ικανοποιεί κάποιες ε, απαιτήσει ε, βιωσιμότητας και υπάρχουν και δείκτες σε ό,τι αφορά το γαλακτοκομικό κλάδο. Και οι γαλακτοκομικές λοιπόν εκμεταλλεύσεις έχουν ε, απευθυνθεί σε ενώσεις, σε συνεταιρισμούς, γιατί τους ενδιαφέρει προφανώς. Αν μας επιτρέπει αυτό να κάνουμε επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων και να τα επισημαίνουμε με τις ετικέτες μας, μας ενδιαφέρει. Άρα υπάρχουν δύο πτυχές. Αφενός μπορούμε να δώσουμε νέες ευκαιρίες για να ενσωματώσουμε στην ετικέτα του προϊόντος τον τρόπο παραγωγής, προκειμένου να ξέρει ο καταναλωτής τι καταναλώνει, τι αγοράζει, τι πληρώνει, κατά πόσο πρόκειται για βιώσιμο προϊόν. Και από την άλλη, σε κάποιες περιπτώσεις θα αυξηθεί το κόστος ε, παραγωγής και δεν θα είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί. Ουσιαστικά η γεωργία παρέχει υπηρεσίε τις οποίες ως κοινωνία α, ε, θεωρεί σημαντικές. Άρα θα πρέπει να δοθεί ε, επιβράβευση, αποζημίωση στους αγρότες και με άλλον τρόπο για αυτό το δημόσιο αγαθό. Αυτό θα μπορούσε λοιπόν να ε, περιλαμβάνει και υποστήριξη σε αποκεντρωμένες περιοχέ. Ε, όπου παρέχονται κάποιες υπηρεσίε οι οποίες αλλιώ θα εκλείπαν. Να υπάρχει σαφέστερη λοιπόν σύνδεση. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν πιο εφικτός τρόπος. Αυτό είναι το πολιτικό συγκείμενο στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν το σκέλος αυτό. Ε, παραμένει και μία τελευταία ερώτηση. Έχετε το λόγο. Δεν άκουσα την απάντηση στην ερώτησή μου θα ήθελα εσείς ως ερευνητές να μου πείτε ποιο είναι το ευεργέτημα για την κοινωνία από μια αγροτική πολιτική η οποία δεν εγγυάται μια ε, σωστή ε, πληρωμή των αγροτών για την ε, εργασία τους μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου. Γιατί θα πρέπει να καταβάλει η κοινωνία φόρους, να βγαίνει το, το χρήμα από το δημόσιο φορέα. Θα ήθελα μία απάντηση να μου πείτε γιατί αυτή η φτηνή πρώτη ύλη. Λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, εάν μπορείτε, με βάση τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας. Και τώρα σε σχέση με τις... και φυσικά και σχέση με τις μελέτες στις διάφορες χώρες, εάν τα έχετε αυτά τα στοιχεία. Ακούστε, σε κάποιο βαθμό πρόκειται για πάρα πολύ βασικό θεμελιώδες ερώτημα, πολύ καλό, αλλά δεν καλύπτεται από το πεδίο της μελέτης που είχαμε συγκεκριμένους στόχους. Ε, οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Ε, σίγουρα έχετε ε, αναφερθεί και εσείς ορισμένα στοιχεία, αλλά αυτά που λέτε δεν ήταν το βασικό αντικείμενο της μελέτης μας, δυστυχώς, οφείλω να το πω. Αλλά για να απαντήσω το ερώτημά σας, θα έπρεπε να συγκρίνουμε ουσιαστικά το πραγματικό κόστος ε, τροφίμων με συγκριτικό τρόπο και να δούμε πώς ε, καλύπτεται, πώς πληρώνεται. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά θα ήταν μια άλλη μελέτη αυτή, αν θέλαμε κυρίω να το κάνουμε σωστά. Και για την πραγματική τιμή και τα σχετικά, το true pricing, ε, νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα, αλλά η μεθοδολογία από την άλλη δεν είναι και τόσο έγκυρη ακόμη, ώστε ε, να μην υπάρχουν προβλήματα. Κάποιες φορές έχουμε προβλήματα, δηλαδή στις συγκρίσεις, γιατί η μεθοδολογία δεν είναι αρκετά παγιωμένη, πώς να το πω. Πρόεδρος, νομίζω ότι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο για τις πληροφορίες ε, τις οποίες ε, μοιραστήκατε μαζί μας. Έχουμε επομένω στη διάθεσή μας τώρα παραπάνω επιχειρήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε την κοινή γεωργική πολιτική, να την υπερασπιστούμε. Βέβαια, Μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική, να βες και από αμφισβήτηση ε, τη, μέχρι τώρα λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, διότι πρέπει να διερωτηθούμε τελικά ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε. Γνωρίζουμε ότι το μερίδιο της κοινή κοινωνικής πολιτικής ε, έχει μειωθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης και θα μειώνεται όλο και περισσότερο. Όμως, παρόλα αυτά, είναι σημαντική η πολιτική αυτή. Κάτι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον επίσης και να λάβουμε επίσης υπόψη μας ότι όταν ακριβένουν τα πάντα, τι γίνεται τελικά και με τη Γεωργία. Αυτή είναι μια σημαντική απορία έτσι. Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε στις 18 και 19. Φεβρουαρίου και 27 Φεβρουαρίου και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. σε σχέση με όσα έχουν απομείνει να διευθετήσουμε μέχρι το τέλο τη θητεία και δείτε η μετάσχεση τη γεωργική πολιτική. Αυτά δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιε παρατηρήσει από του βουλευτέ. Αν όχι, Επιτρέψτε μου να κηρύξω τη λήξη συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε. Ευχαριστώ και του διερμηνεί ο πρόεδρο.